επαναλαμβάνονται συνεδρίαση και τα πρακτικά της θεσινής συνεδρίασης έχουν διανεμηθεί. Αν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, ε, θεωρείται πως τα πρακτικά εγκρίνονται. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, θα συζητήσουμε την έκθεση του κυρίου Φρανσίσκου Χωσέ Μιλαμόν για την κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων την επαύριο των εκλογών στις ΗΠΑ. Το λόγο έχει ο εισηγητής κύριος Μίλαν Παρακαλώ. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τους χιώδες εισηγητές, κύριε συγκεκριμένα Σαβαρή, Λάμπστορφ και επίσης Γαρθία Μαργάγιο και Κίστεν Ρόμπολ που έχουν συντάξει κάποιες γνωμοδοτήσεις με βοήθησαν πάρα πολύ ούτως ώστε να μπορέσουμε να συντάξουμε αυτή την έκθεση για